κατοίκων του Νεπάλ. Εμείς βεβαίως και θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και θα προετοιμάσουμε νέα έκθεση στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Τέλος της συζήτησης και βεβαίως θα ψηφίσουμε ακριβώς μετά το τέλος του τελευταίου κατεπήγοντος θέματος που είναι η κατάσταση στην Ζιμπάμπουε. Δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Πρόεδρε, που ασχολούμαστε με τα τεκτενόμενα στην Ζιμπάμπουε, με το κόμμα του Γκάμπε και το καθεστώς αυτό το οποίο συνεχίζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ζιμπάμπουε. Πρόκειται για συλλήψεις, για εξαφανίσεις, για διωγμούς των πολιτικών αντιπάλων. Τα πολιτικά κόμματα φοβούνται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουν με έναν ε, κανονικό εκλογικό με μια κανονική ε, και ομαλή εκλογική αναμέτρηση να φτάσουν στην εξουσία. Πολλοί φοβούνται ότι όλα τα μέτρα που έχουν ε, ληφθεί μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από αλλού στον κόσμο για να απελευθερωθούν οι συλληφθέντες δεν έχουν απολύτως κανένα αποτέλεσμα. Η κυβέρνηση Μουγκάμπε συνεχίζει παρόλα αυτά να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να καταδιώκει τον λαό της Ζιμπάμπουε. Σήμερα βλέπουμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται και δεν ακολουθεί το παράδειγμα της Νότιας Αφρικής. Uh, Κύριε Βαν είμαι 12 χρόνια στο Κοινοβούλιο και από τότε που είμαι εδώ προσπαθούμε να βοηθήσουμε το λαό της Ζυμπάγου να ζήσουν καλύτερα, να είναι πιο αισιόδοξοι για το μέλλον που τους περιμένει. Και νομίζω ότι για δύο σημεία έχουμε εκφραστεί πάντοτε με σαφήνεια. Πρώτα απ' όλα το όσο είναι στην κυβέρνηση ο Ρόμπερτ Μουμπά, Μουγκάμπε ε, με την υποστήριξη ε, από τις δυνάμεις ε, επιβολής του νόμου και από το κόμμα του με σκοπό τον προσωπικό πληθυσμό δεν υπήρχε δυνατότητα μεταρρύθμισης και αλλαγής. Και δεύτερον, πως ήταν ο λαός της Ζιμπάμπουε με τη στήριξη των γειτονικών του χωρών και κυρίως Νοτιοαφρικής που θα έπρεπε να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές. Και μόνο τότε θα γινόταν κάποια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Ίσως να έφτασε η στιγμή. Ξέρουμε πως όταν ανησυχεί ο Μουγκάβε αρχίζει να πανικοβάλλεται. Η αστυνομία και οι παραστρατιωτικές δυνάμεις επιτίθενται σε όποιον θεωρούν εχθρό. Η MDC υποτίθεται πως είναι σε συνασπισμό μαζί τους, αλλά τις τελευταίες μέρες οι βουλευτές αυτού του κόμματος, οι ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και οι υπουργοί έχουν ξυλοκοπηθεί και συλληφθεί γιατί ο Ρόμπερτ Μουγκάβε ανησυχεί. Ανησυχεί γιατί βλέπει τι πάθαν οι φίλοι του. Και κυρίω ο βασικό του χρηματοδότη ο Καντάφη. Και στι 31 Μαρτίου, πριν μια εβδομάδα, είχαμε την ε, κοινότητα ανάπτυξη Νοτιοαφρικής με όλους τους γείτονες της Νοτιοαφρικής και της Ζιμπάμπουε εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία επιτέλους για την αύξηση της βίας στην Ζιμπάμπουε και ζήτησε ε, η πολιτική συμφωνία, η, συνολική, σφαιρική πολιτική συμφωνία να εφαρμοστεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης για να γίνουν δίκαιες και ελεύθερες εκλογές στη Ζιμπάμπουε. Και σήμερα αυτό γίνεται στην Χαράρε ε, ζητάμε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εντοκοποιήσουν τη συμμετοχή τους και να χρησιμοποιήσουν όλη τους την πολιτική επιρροή στη Νότια Αφρική για να γίνει μια κίνηση προς τα εμπρός, μια βελτίωση της καταστάσεως και μια παρατήρηση των εκλογών έτσι ώστε να γίνουν αυτές με ελεύθερο τρόπο. Όντως βλέπουμε φαινόμενα αλλαγής και τα μέτρα τα οποία ισχύουν κατά του Μουγκάβη και των στενών του συμμάχων θα πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους. δεν θα πρέπει εμείς ε, να θεωρήσουμε πως ο μονομερός διορισμένος, απεσταλμένος του ε, Ζιμπάμπου είναι πρέσβης εδώ σε εμά. Όταν λοιπόν εγκατασταθεί το κράτος δικαίου στη Ζιμπάμπου είμαι σίγουρος πως η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει γενναιόδρα τη χώρα αυτή να σταθεί στα πόδια της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βανόδεν. Η κυρία Σαργεντίνη. Ευχαριστώ. Εδώ και δέκα χρόνια ασχολούμαι με την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε, με αναπτυξιακές οργανώσεις στο Άμστερνταμ, με ακτιβιστές στην Ολλανδία και στην Ευρώπη. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, να ακούσουμε τις ιστορίες αυτών των ε, ανθρώπων που έχουν διωχθεί. Μιλήσαμε στο ψήφισμα για την περίπτωση Γουσικόμου. Είναι ένας ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος ήταν ενθουσιώδης και ο οποίος ε, δεν έχει χάσει τον ενθουσιασμό του. Σε τέτοιους ανθρώπους απευθυνόμαστε με αυτό το ψήφισμα. Δεν ξέρω ότι ο κύριος ε, Μουγκάμπε χάνει τον ύπνο του. Οι συνάδελφοι, οι πολιτικοί του MDC θέλουν να συνεχίσουν με τη δική τους ατζέντα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σε σχέση με τις κυρώσεις. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ισχύ της διαδικασίας Κίμπερλι δηλαδή να ισχύσει η σωστή διαδικασία στα αδαμαντορυχεία και τη στιγμή που δεν πληρούνται οι όροι να μην πολλούνται, να μην μπορούν να πολιθούν αυτά τα διαμάντια γιατί αφορούν ακόμα και παιδική εργασία. Πολλές φορές ε, θα πρέπει να αναφερόμαστε, συνεχώς θα πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτούς τους ε, θαραλέους ανθρώπους. Οίλαντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ανησυχώ με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ζιμπάμπουε που επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες. Και αυτή η ανησυχία βεβαίως φαίνεται από τις νέες εντολές που δόθηκαν στην χώρα αυτή. Η αντιπολίτευση, η πολιτικοί και οι ακτιβιστές οι οποίοι έχουν συλληφθεί, έχουν βασανιστεί και περιοριστικά μέτρα για την ελευθερία των πολιτών έχουν επιβληθεί από το καθεστώς Μουγκάμπε και βεβαίως μέχρι να υπάρξει απόδειξη ότι αλλάζει το καθεστώς η κατάσταση είναι ανησυχητική. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες της χώρας αυτής να μπορούν να εκφραστούν χωρίς να φοβούνται συλλήψεις, βασανισμούς και η κυβέρνηση αυτή θα πρέπει να κατηγορηθεί και να προσταθεί. Η καταστολή στη Ζιμπάμπουε αποτελεί ε, ένα σαφές μήνυμα για τις ε, επόμενες εκλογές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οργανώσεις όπως η ΣΑΔΚ, η Κοινότητα για την Ανάπτυξη Μεσημβρής Αφρικής, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη να μην καταδιώκονται, μην διώκονται ακτιβιστές του ΕΜΤΕΣΕ πριν από τη διενέργεια εκλογών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις εισβολές που γίνονται στα γραφεία ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να βρεθεί δήθεν ανατρεπτικό υλικό. Αυτό αφορά και τους φοιτητές ακτιβιστές. Πρόκειται για τακτική μίας εκστρατείας εκφοβισμού που είναι απαράδεκτη. Επίσης γίνεται εκφοβισμός κατά εκείνων που ε, δεν υπογράφουν την άρση των ε, περιοριστικών μέτρων. Όλα αυτά έχουν σχέση με την άνοιξη του αραβικού κόσμου, που βεβαίως θα έχει μεγάλη επιρροή σε αυτή την περιοχή. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι μιλώ από πλευράς ε, του συναδέλφου Αλκαντέκ, ο οποίος δεν είναι εδώ το απόγευμα. Αυτά τα τρία θέματα, από αυτά τα τρία θέματα, αυτό είναι ένα θέμα που ανακύπτει όλο ένα και περισσότερο. Ο Μουγκάμπε έχει κυβερνήσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με μεγάλη βιαιότητα σε αυτή την χώρα. Και η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας το 2009 που υποτίθεται ότι θα έφερνε τη δημοκρατία δεν είναι λειτουργική. Δυστυχώς, τους τελευταίους μήνες με την εκστρατεία εκφοβισμού, τις συλλήψεις και τις εξαφανίσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι κατασταλτικά μέτρα τα οποία είναι απαράδεκτα. Ακόμα και οι μη κυβερνητικέ έχουν αποτελέσει αντικείμενο αυτής της εκστρατείας εκφοβισμού θα πρέπει να σταματήσουμε τη δράση αυτού του δικτάτορα. Και τώρα η, η Αφρικανική Ενότητα δημιουργεί ένα συνασπισμό κατά του Μουγκάμπε και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να συνταχθούμε με εκείνους και να καταβάλουμε κάθε διπλωματική προσπάθεια που έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε ο κύριος Μουγκάμπε να σταματήσει τις συλλήψεις και τις εκτελέσεις, να γίνει αποδεκτό το Σύνταγμα και μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος των βασικών ελευθεριών για να φτάσουμε στην διενέργεια ελευθέρων εκλογών και δημοκρατικής κυβέρνησης στη Ζιμπάμπουε. Ο κύριος Σταβάρες έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όλοι γνωρίζουμε ότι η συμφωνία του 2008 που τέθηκε σε ε, εφαρμογή το 2009 μεταξύ Ζάνου και MTC δεν ήταν μια, ε, ένα σωστό συνασπισμός μεταξύ Μουγκάμπε και Τσβάνγκυράι. Είναι γεγονός ότι ο Μουγκάμπε και οι σύμμαχοί του κατέβαλαν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να μην λειτουργήσει αυτή η συμφωνία. Έγινε μεγάλη εκστρατεία εκφοβισμού, κατεστάλη η αντιπολίτευση που πλειοψηφεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Όλα αυτά έγιναν γνωστά. Πολλές επιθέσεις κατά πολιτών και διαδηλώσεων από το MDC. Εμείς παρακολουθούμε την κατάσταση εκ του σύνεγγης. Δεν θα πρέπει να δεχτούμε αυτό το, αυτή τη νέα παγίδα, το τέχνασμα του Μουγκάμπε που όρισε μία νέα πρέσβυρα χωρίς, χωρίς τις σωστές ε, προεργασίες διαπιστευτηρίων. Δεν θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές αυτές οι καταστάσεις. Τώρα, εξ των πολιτικών ομάδων, Κατσμάρεκ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω πως η κατάσταση στη είναι εξαιρετικά ανισχύ και μάλιστα τώρα που εορτάζεται η επέτειος απελευθερώσης της χώρας. Λοιπόν, τα στοιχεία που μας απασχολούν είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί τα προβλήματα της Ζιμπάμπου είναι πάρα πολλά. Είναι μια χώρα που οι νόμοι δεν αποτελούν προϊόν της δημοκρατικής απόφασης των πολιτών, αλλά επιβάλλονται από μια δικτατορία. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ζητήσουμε να γίνουν σεβαστές μια σειρά από προϋποθέσεις. Καταρχήν, ανθρώπινα δικαιώματα, βελτίωση στον κλάδο αυτό και γι' αυτό ε, το θίγω εδώ, γιατί μπορεί κανείς να αμφιβάλλει για το κατά πόσο τα κατασταλτικά αυτά μέτρα είναι σωστά και αν, με συγχωρείτε, τα διάφορα εμπάργκο που έχουν επιβληθεί είναι και τα περιοριστικά μέτρα λειτουργούν σωστά ή όχι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό γιατί αυτό που συμβαίνει στην ε, Ζιμπάμπου είναι ότι όσοι ζητούν ανθρώπινα δικαιώματα ξυλοκοπούνται και φυλακίζονται. Ο μέρος των σοσιαλιστών είναι ο κύριος Αρσένης το κόμμα του Μουγκάμπε και οι μηχανισμοί του αυτή τη στιγμή, όπως είπαν οι συνάδελφοι, απειλούν, βασανίζουν, χτυπούν οποιονδήποτε αγωνίζεται για τη δημοκρατία και τις δημοκρατικές ελευθερίες στην, ε, στην χώρα, στη Ζιμπάμπουε και τη μετάβαση σε ένα ομαλό δημοκρατικό καθεστώς. Έχουμε ευθύνη για το τι γίνεται στην Αφρική. Στην ιστορία της, το, της δημοκρατίας στην Αφρική έχουμε παρέμβει πάρα πολλέ φορέ ιδίω στην αρχή τη δημιουργία αυτών των νέων χωρών ε, έχουμε εμποδίσει δημοκρατικέ διαδικασίε όταν απειλούνται και τα δικά μα συμφέροντα. έχουμε οπότε διπλό χρέο να βοηθήσουμε να αποκτήσει η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. συναισθηματικά αυτή η κατάσταση για τους έλληνες είναι ιδιαίτερα σημαντική. το 1967 με 74 είχαμε μια πάρα πολύ σκληρή δικτατορία και τότε οποιαδήποτε καταδίκη ερχόταν από το συμβούλιο της ευρώπης ή διεθνούς οργανισμούς έδινε μια ελπίδα σε όλους τους πολίτες που αγωνίζονταν στην ελλάδα. γι' αυτό το λόγο πρέπει να μην δεχτούμε οποιαδήποτε σχέση με παράτυπα διορισμένους εκπροσώπους της ζιμπάμπουε και τους πρώην συνεργάτες του καθεστώτος μουγκάμπε και πρέπει να εγγυηθεί η ευρωπαϊκή ένωση μαζί με τις χώρες της περιοχής τη μετάβαση της ζιμπάμπουε στην δημοκρατία αλλά και την εφαρμογή της διαδικασίας κίμπερλι. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τανόκ, επόμενος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη διαδικασία του Κίμπερλι που έχει ως σκοπό να, ξε περαστούν οι σειράξει και να εξαφανιστούν τα διαμάντια του αίματο από την παγκόσμια αγορά. Όμω οι εξελίξει επόμενα είναι σχετικέ. Ο κύριο Μάθιο Γιάμπα από το Κονγκό, που είναι πρόεδρο αυτή τη διαδικασία, μονομερό και χωρί διαβούλευση, επέτρεψε την θέση σε εμπορία διαμάντα από το ρηχείο Μιράγκη στην Ζιμπάμπουε, το οποίο πέρσι άρπαξαν ο πρόεδρο Μουγκάμπε και οι φίλοι του, έδιωξε εκατοντάδε ανθρώπου από, από τα σπίτια του, και είχαν ε, σημειωθεί κρούσματα βασανιστήριων, αρπαγών, ε, ε, ως και φόνων ανθρώπων που δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αυτό έγινε για να πλουτίσει ο κύριος Μουγκάβε και το κόμμα του. Ζητώ λοιπόν το σκάνδαλο αυτό να το θέσει στην κορυφή της ατζέντα, στα πλαίσια της διαδικασίας του Κίμπερλι, έτσι ώστε να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο λήψης αποφάσεων μέσα στη διαδικασία του Κίμπερλι. Πρέπει να καλύψουμε και τα άλλα τις άλλες πρώτες που εξορίσονται στην Αφρική έτσι ώστε να αυτές οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις να μην πουλάνε πολύτιμες πρώτες ύλες για να αγοράζουν όπλα. Εγώ συνεργάζομαι με την Global Witness που είναι πολύ γνωστή με στο θέμα αυτό και η πράξη Dodd Frank στι ΗΠΑ πραγματικά μας δείχνει το δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπρέντα είναι ο επόμενο Ευχαριστώ πολύ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση Ζιμπάμπου που μας θυμίζει το καθεστώς του Νικολάη Τσαουσέσκου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Καντάφη ήταν μεγάλος φίλος του Τσαουσέσκου κατά τη δεκαετία του 80. Και η κατάσταση αυτή δείχνουν, δείχνει και τη σχέση Μουγκάμπε-Καντάφη. Όμως ο Μουγκάμπε έμαθε, πήρε πολλά μαθήματα από, από τον Τσαουσέσκου και ε, συνέλαβε πολλούς ακτιβιστές και μέλη κοινωνίας των πολιτών. Θα φυλακιστούν και θα καταδικαστούν στη θανατική ποινή το μόνο τους αμάρτημα είναι ότι συζήτησαν για το τι έγινε στην Αίγυπτο και την Τινησία. Θα πρέπει να διενεργηθούν ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές στη Ζιμπάμπουε και ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μασάια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ψήφισμα για την Ζιμπάμπουε λέγοντας ότι θα πρέπει να παραμείνουν οι κυρώσεις καθότι δεν βλέπουμε σημαντική πρόοδο όπως είχαμε ζητήσει πραγματική πρόοδο όσον αφορά την συμφωνία για την συμμετοχή στην εξουσία των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Η δυνάμεις ασφαλείας, ιδιοκτικές αρχές βασανίζουν, δολοφονούν, συλλαμβάνουν τους αντιφρονούντες και την αντιπολίτευση. Και πολλές φορές βλέπουμε τα εγκλήματα αυτά να διαπράττονται κατά απλών πολιτών της Ζιμπάμπουε. Υπάρχουν προβλήματα με τους φυσικούς πόρους και πιστεύω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να στείλουμε παρατηρητές κατά τη διάρκεια των εκλογών. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι η τελευταία συζήτηση που έγινε για την Ζιμπάμπουα ήταν πέρα και από τότε μέχρι σήμερα Τίποτα απολύτως δεν έχει αλλάξει. Υπάρχει 90% ανεργία, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν υπάρχει πρόσβαση αυτών που ζουν στην επαρχία σε βασικές υπηρεσίες και βλέπουμε πολύ καλά ότι η συμφωνία μεταξύ Μουγκάμπε και Ζαγκύρα δεν πληρεί καμία από τις απαιτήσει και τους στόχους η κατάσταση εκτός της χώρας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Βλέπουμε σήμερα τι γίνεται στη Βόρεια Αφρική. Κάποια χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίζουν βεβαίως την Βόρεια Αφρική και την Ζιμπάμπουε. Βλέπετε όμως τι γίνεται και στην ακτή του Ελεφαντοστούν σήμερα. Καταρχήν λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να εμποδίσουμε περαιτέρω σύλληψεις και διώξεις της αντιπολίτευσης. Η Ζιμπάμπουε δεν μπορεί πλέον να δημιουργεί τεχνητά προβλήματα, αλλά να, λύσει τα πραγματικά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Πούσεκ. Ευχαριστώ πολύ. Ως μέλος της αντιπροσωπείας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με, το, ε, με την Παναφρικανική Ένωση θεωρώ ότι η κυρία Άστον θα πρέπει να στραφεί κατά αυτών των δράσεων εκφοβισμού της κυβέρνησης ε, Μουγκάμπε και θα πρέπει να τηρηθούν οι βασικές ελευθερίες, η ελευθερία του λόγου και του συνέρχεστε η Ζιμπάμπουε θα πρέπει να δεχτεί τις διεθνείς συμφωνίες όπως και τον Αφρικανικό χάρτη και να καταργήσει κάθε εθνικό νόμο που δεν δέχεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρώ ότι η Νότιος Αφρική θα μπορούσε να υποστηρίσει τη, διαδικασία ε, ε, πανισδοχής της Ζιμπάμπουε στο δημοκρατικό κόσμο. Η κυρία Μπασέσκου έχει το λόγο. Στα ρουμανικά. Εκ νέου. Βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολύ μεγάλη απειλή καταστολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το, από τον Ιούνιο και μετά ο πρόεδρος Γκάμπε προσπαθεί να εκφοβήσει όλους τους υποψηφίους. Επίσης, πολλά μέλη της αντιπολίτευσης έχουν φυλακιστεί και συλληφθεί τους τελευταίους δύο μήνες. Θα πρέπει να καταρτιστεί ένα νέο σύνταγμα, το οποίο όμως έχει ανασταλεί εδώ και ένα χρόνο από την κυβέρνηση Μουγκάμπε. Θα πρέπει να υπάρχουν συνθήκες διαφάνειας και να μην ξεχνάμε ότι στη χώρα αυτή υπάρχει μεγάλος σκοτάδισμος. Επίσης, δεν μπορεί να ισχύσει η διαδικασία Κίμπερλι για τα αδαμαντορυχεία. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την οικονομική ε, κατάσταση. Το λόγο έχει ο κύριος... Ε, ο κύριος Ρέπο, ευχαριστώ πολύ. Το κόμμα του κυρίου Μουγκάμπε δεν σεβάστηκε τη συμφωνία για το επιμερισμό της εξουσίας και δεν κατάφερε να κάνει τη μετάβαση προς τη δημοκρατία η Ζιμπάπουε. Αυτή τη στιγμή κυριαρχεί ο φόβος, οι συλλήψεις, τα βασανιστήρια και όλα αυτά αυξάνονται τους τελευταίους μήνες. Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπει να σημειωθεί πρόοδος και βασανίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις, ε, για παράδειγμα δημοσιογράφοι, οι οποίοι έχουν υποστεί βασανιστήρια για το όσα έγραψαν. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τη Ζιμπάμπουε σε επίπεδο αναπτυξιακό και νομίζω πως η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αποφάσισε να συνεχίσει με τα περιοριστικά μέτρα ε, που έχει επιβάλει στην ε, κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε με το γνωστό κατάλογο ε, είναι εξαιρετική γιατί πρέπει να δούμε πρώτα πως όντως γίνονται κάποιες μεταρρυθμίσεις στην Ζιμπάμπουε πριν άρουμε τα μέτρα αυτά. Θα πρέπει όμως τα μέτρα αυτά να εστιάζονται στα κυβερνητικά στελέχη και όχι γενικότερα στο λαό της Ζιμπάμπουε. Και τελευταία ομιλήτρια. Ζητήσατε το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ μικρό παιδί είχα πάει στην Ροδεσία και θυμάμαι ότι ήδη από τότε υπήρχε λογοτεχνία για τις περιοχές αυτές, για την Νότια Αφρική και την τότε Ροδεσία. Η κατάσταση σήμερα είναι απαράδεκτη. Η Ροδεσία που σήμερα ονομάζεται Ζιμπάμπουε βρίσκεται υπό την κατοχή του Μπουγκάμπε. Ο κόσμος υποφέρει από πείνα και από διάφορες διώξεις και πραγματικά Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους συναδέλφους που έφεραν το θέμα αυτό στην επικαιρότητα γιατί είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει στην χώρα αυτή. Πρόκειται για ένα δικτατορικό καθεστώς και όσο η Νότια Αφρική δεν κάνει κάτι έτσι ώστε να εξαφανιστεί αυτός ο δικτάτορας δεν θα μπορέσουν οι πιέσεις να κάνουν απολύτως τίποτα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα ζητήσω από τον κύριο Σεύκοβιτς από την Επιτροπή να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι έχουμε ανοιχτεί αυτές παραβιάσεις και το θέμα αυτό είναι εδώ και πολύ καιρό στην ημερήσια διάταξη. Και κάθε φορά που υπάρχει μια αισιοδοξία και ένα θετικό γεγονός αυτό εξαφανίζεται από ένα κύμα, κάτω από ένα κύμα διώξεων και παραβιάσεων. Πιστεύω πραγματικά ότι θα πρέπει να δούμε αυτά που έγιναν το Φεβρουάριο του 2011, παραδείγματο χάρη. Είναι σαφές ότι η συμφωνία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης έχει μεγάλη σημασία. Φαίνεται ότι υπάρχει βούληση να αναθεωρηθεί η απόφαση που έχει ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν υπάρξουν θετικές εξελίξεις επιτόπου. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τα τελευταία γεγονότα. Τον Μάρτιο με πολλές ε, πρεσβείες επιτόπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει την ανησυχία της όσον αφορά τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις διώξεις, συλλήψεις και την βία στην χώρα αυτή. Στις 31 Μαρτίου του 2011 υπήρξε η ανακοίνωση για τις ε, βίες πράξεις, τις συλλήψεις, τις διώξεις που λαμβάνουν χώρα στη χώρα αυτή και οι οποίες θα πρέπει να πάψουν αμέσως. Εν ώψη των ε, εκλογών που διοργανώνονται, θα πρέπει να βοηθήσουμε με ειδικούς, με παρατηρητές, οι οποίοι θα συνεργαστούν με την ομάδα από την Νότια Αφρική, για να αποφύγουμε περαιτέρω αστάθεια και βία στην Ζιμπάγκουε και περαιτέρω πολιτική κρίση. Η Νότια Αφρική μπορεί να παίξει εδώ ένα ρόλο μεσολαβητή έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια γενικότερη συμφωνία επιτόπου. Συνεχίζουμε βεβαίως να έχουμε κανάλια επικοινωνίας με την Ζιμπάμπουε και διάλογο με την κυβέρνηση γιατί δεν θέλουμε να εξασθενήσουμε τη θέση μας επιτόπου η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο πρώτος χορηγός βοήθειας στην Ζιμπάμπουε. Προσπαθούμε να μην στηρίξουμε την δικτατορική κυβέρνηση, αλλά τον λαό της Ζιμπάμπουε. Και προσπαθούμε μέσω μιας συνολικής συμφωνίας να βοηθήσουμε τους φυσικούς πόρους οι οποίοι διοχετεύονται και χορηγούνται μόνο μέσω μη κυβερνητικών οργανισμών μέχρι να υπάρξει μια γενικότερη πολιτική συμφωνία και συνταγματική μεταρρύθμιση. Επίσης στηρίζουμε τους ε, ανθρώπους επιτόπου οι οποίοι προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και προσπαθούν να στηρίξουν την διοργάνωση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, παρόλο που η κατάσταση συνεχίζει να μας ανησυχεί και να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Επίτροπε, η συζήτηση για τη Τζιμπάγκου, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει λήξει και μπορούμε να ψηφίσουμε. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη ψηφοφορία για τον Ai Weiwei. Έχουμε έξι προτάσεις ψηφισμάτων τροπολογία